Σας ευχαριστώ. Τελείωσε η συζήτηση. Η ψηφοφορία επίσης αύριο στις 12. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Την έκθεση του κυρίου Γουίντο Μιλάνα για την στρατηγική για την αλληλεία στην Αδριατική και στο Ιόνιο. Και εσύ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της, διότι ε, μπορέσαμε της Επιτροπής μας, συγγνώμη, της Επιτροπής η οποία ενέκρινε την πρόταση αυτή με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και ελπίζω να είναι αντίστοιχη ψηφοφορία αύριο στην Ολομέλεια, διότι έτσι θα έχουμε... Ε, καλές δυνατότητες για τους αλληλεί της Αντιρατική θάλασσας και του Ιωνίου Πελάγους, αλλά ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να έχουμε και το εναρκτήριο λάκτισμα για την κατάλληλη πολιτική για τη Μεσόγειο. Καταρχάς λοιπόν να σας ε, παρουσιάσω λίγο το πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια συγκεκριμένη θαλάσσια πολιτική για την Αδριατική θάλασσα. Έχει φτάσει πλέον η στιγμή, αυτό ορίμασε με την ανακοίνωση που έγινε πέρσι ε, κατόπιν όθησης ε, των χωρών της Αδριατικής, ε, της Ιταλίας, της Κροατίας που μόλις εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίστηκε η ανάγκη να υπάρχει μια συνολική θαλάσσια πολιτική στην περιοχή αυτή και εδώ εντάσσεται και η συγκεκριμένη έκθεση. Διότι στην ουσία καλύπτει κάποιες από τις ιδιαιτερότητες αυτής της θάλασσας. Ένα άλλο σημαντικό πλαίσιο ε, στο οποίο εμπίπτει αυτή η τόσο σημαντική έκθεση που θα εγκρίνει αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετίζεται με το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει πλέον η νέα αλλιευτική πολιτική. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει την μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής ε, πολιτικής εντός ε, του έτους και φυσικά θα υπάρχει και χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλείας ώστε να καθοριστούν οι πόροι για την ανάπτυξη του τομέα αυτά στα επόμενα χρόνια. Και αυτό λοιπόν είναι σημαντικό διότι η έκθεση συμβαίνει σε μια κέρια χρονική στιγμή κατέστη σαφές ότι η παρούσα νομοθεσία στη συγκεκριμένη θάλασσα είναι πολύ γενικόλογη και δεν μπορεί να ρυθμίσει συνολικά τα προβλήματα της συγκεκριμένη ε, περιοχής. Η Αδριατική θάλασσα, σε αντίθεση με τη Μεσόγειο, είναι μια κλειστή θάλασσα, είναι μια θάλασσα στην οποία συνεπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι εντελώς διαφορετικού οικονομικού χαρακτήρα σε σχέση με την υπόλοιπη Μεσόγειο υπάρχουν διαφορετικά, ε, διαφορετική ποικιλία στο βυθό, είναι τελείως διαφορετική η αλληλευτική παράδοση και ε, η, τα διεθνή ύδατα είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με την υπόλοιπη Μεσόγειο. Έχουμε μια κλειστή θάλασσα με τρεις χώρες οι οποίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιταλία, Σλοβενία και Κροατία και τρεις άλλες χώρες οι οποίες έχουν τελείως διαφορετική πολιτική, άλλη νομοθεσία και άλλους μηχανισμούς. Και απ' την άλλη είναι τόσο κοντά και τόσο αλληλένδεδες αυτές οι χώρες. Και σε αυτές τις χώρες υπάρχει η ίδια νομοθεσία με την υπόλοιπη Μεσόγειο. Και αυτό φυσικά δημιουργεί προβλήματα γιατί οποιαδήποτε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει να γίνει μάταιη. Είναι μάταιος ο έλεγχος ε, στις θάλασσες αυτές, ακόμα και αποτελεσματικότητα για την προστασία των αποθεμάτων. Και ουσιαστικά η αλληλεία πτωχεύει και ορισμένες φορές αποτελεί οικονομικό και κοινωνικό βάρος και μάλιστα δυσβάσταχτο. Η Επιτροπή λοιπόν Αλίας ε, και ελπίζω αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσαν τις κατάλληλες καταυθυντήριες γραμμές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει υπόψη της δύο σημαντικά στοιχεία. Ένα νέο πρόγραμμα δράσης το οποίο θα είναι εκ διαμέτρου αντίθετο και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα συνύπαρξης κοινοτικών και μη κοινοτικών χωρών σε μια τόσο κοντινή περιοχή αυτή τη στιγμή που ξεκινάει η μεταρρύθμιση και δεύτερον το γεγονό ότι δεν μπορούμε να έχουμε γενικούς κανόνες για όλη την Ευρώπη διότι υπάρχουν αντικειμενικές διαφορές. Και αυτό φυσικά ε, καλύπτεται από μια ιδιαίτερη συζήτηση η οποία προκύπτει στο συγκεκριμένο τομέα της ε, ε, περιφερειοποίησης. Αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε γενικούς κανόνες αλλά με τοπική εφαρμογή θεωρώ ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό λιθαράκι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τέσσερις ομιλητές έχουν στήσει το λόγο κύριος Μπλέγκοβιτς είναι πρώτος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Μιλάνα, για τις προσπάθειές του. Και βεβαίω το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για εμάς στην Κροατία και θεωρώ πως μια συνολική στρατηγική θα βοηθήσει τους αλληλείς σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τις θάλασσες αυτές ειδικά όσους θέλουν να τηρήσουν τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η αλληλείς ε, στην Κροατία. Νομίζω πως η αλληλεία πρέπει να είναι βασική οικονομική δραστηριότητα στον τομέα αυτών και σας απευθύνω έκκληση να δώσετε ιδιαίτερο βάρος στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. Ειδικά στις προσπάθειες ε, για να, για να αποτραπεί η εγκατάλειψη των νησιών αυτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή και να σημειώσω πως ε, ε, πω όταν ε, συνταχθεί η έκθεση έχει ενταχθεί η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί εδώ πέρα αναφέρεται πως θα ενταχθεί. Πράγματι, σωστά αναφέρονται κάποια προβλήματα στη συνεργασία στην Αδριατική και υπάρχουν κάποια τμήματα της Αδριατικής που δεν καλύπτονται από τις οικολογικές και αλευτικές ζώνες. Οι οικολογικές και αλευτικές ζώνες της Κροατίας ισχύουν μόνο για τρίτες χώρες, όχι για τα κράτη-μέλη, αλλά το σημαντικό μήνυμα εδώ πέρα είναι πως το πνεύμα της έκθεσης ε, είναι να εφαρμοστούν όσα ισχύουν ε, στην Κροατία και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα αυτό λοιπόν θα τεθεί μόλις ε, καθοριστούν τα όρια μεταξύ βεβαίως Κροατίας και Σλοβενίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Τόμασικ. Η κυρία Τόμασικ, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα καθότι προέρχομαι από την Κροατία το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προστασία των αποθεμάτων, των αλληλευτικών αποθεμάτων στην περιοχή, για όλες τις χώρες της περιοχής και πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προστασίας έτσι ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν αλληλευτικά αποθέματα. Στηρίζουμε επίσης τις προσπάθειες των παράκτιων περιοχών για μια πιο βιώσιμη και πιο περιβαλλοντολογικά σωστή ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή βεβαίως προϋποθέτει περισσότερο έλεγχο από μέρους των κρατών μελών και περισσότερα μέτρα για την προστασία της Μεσογείου. Η περιοχή της Μεσογείου θα πρέπει να γίνει με τον αποκοινού έλεγχο όλων των ε, χωρών της Μεσογείου, εξετάζοντας βεβαίως και τις επιπτώσεις επί της οικονομίας. Θα vidite ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για μας την Κροατία. Πόσο σημαντική είναι η Αδριατική θάλασσα, η περιοχή της Μεσογείου. Όλοι θέλουμε να πάρουμε το λόγο. Η Κροατία, η Ιταλία και η Ελλάδα βρίσκονται γύρω από την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος και άλλες χώρες βεβαίως όπως η Βοσνία, η Αλβανία έχουν πρόσβαση στην Αδριατική θάλασσα και το Μαυροβούνιο βεβαίως το οποίο είναι υποψήφια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλες χώρες που πολύ θα θέλαμε να συνεργαστούν και να προσχωρήσουν. Χρειάζεται λοιπόν μια συνεργασία και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποθεμάτων και των πόρων μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η καλή διαχείριση της περιοχής αυτής, αυτής της θαλάσσιας ζώνης και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια συμβατή και συντονισμένη προσέγγιση. Στην περιοχή του του υπάρχουν ηχθειοκαλλιέργειες και και καλλιέργειες άλλων ε, θαλάσσιων οργανισμών, την οποία θέλουμε βεβαίω να προστατεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντινγκ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον ε, κύριο Μιλάνα τον εισηγητή. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση και η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία της περιοχής της Αδριατικής θάλασσας και του Ιωνίου. Όλα τα θέματα που άπτονται της θάλασσας, της αλληλείας, της ηχθοκαλλιέργειας, της προστασίας των θαλάσσιων περιοχών βεβαίως περιέχουν και μια τεχνολογική πτυχή, μια πτυχή καινοτομίας. Οι τοπικές αρχές οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να συνεισφέρουν και ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για την επιτυχία αυτής της πολιτικής. Στηρίζουμε λοιπόν αυτή τη στρατηγική έτσι ώστε να υπάρξει και μια συνιστόσα συντονισμού και τα μέτρα τα οποία θα υιοθετούνται να είναι συμβατά με την κοινωτική πολιτική. Θεωρούμε ότι η εκμετάλλευση των ε, πόρων της περιοχής θα πρέπει να βασίζεται σε ίδιους κανόνες, σε κοινούς κανόνες. Η προστασία των ε, αποθεμάτων θα πρέπει επίσης να στηρίζεται στο νέο πλαίσιο συλλογής στοιχείων και δεδομένων. Υπάρχει λοιπόν σήμερα μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα πλαίσιο δράσης το πρώτο εξάμεινο του 2014 για την προστασία αυτών των αποθεμάτων και είναι σαφές από τις προτάσεις της ε, έκθεσης ότι η στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι και το τελευταίο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Είναι η έκθεση Ντελάνγκε, μια περισσότερο αποτελεσματική και